Ε, του συστήματος παρουσίασης ε, δημοσίων εγγράφων. Δίνουμε αμέσως το λόγο στην κυρία Ντελβό. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω από 14 εκατομμύρια πολίτες ζουν σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσης για να ανυμφευθούν, να ανακοινώσουν τη γέννηση του παιδιού τους, να ζητήσουν ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου, υποχρεούνται να υπόκεινται σε διαδικασίες δύσκολες και κοστοβόρες. Δεν αρκεί να καταθέσουν ένα έγγραφο από τη χώρα προέλευσης, πρέπει να συνοδεύεται από μια σφραγίδα η λεγόμενη αποστή της Χάγης. Απαιτείται επίσης και μία εγκεκριμένη μετάφραση. Παρ' όλα αυτά η ελεύθερη διακίνηση είναι ένα βασικό δικαίωμα το οποίο δίδει η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν να γίνει πιο συγκεκριμένο αυτό και αυτό περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα της Στοκόλμης του 2009 για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Δικαιοσύνης προβλέπεται η κατάργηση της αποστήγια. Εφτά χρόνια μετά φτάνουμε και Ο κανονισμός για την απλοποίηση της αποδοχής των δημοσίων εγγράφων είναι ένα βήμα μικρό βέβαια για την ελάφρυνση αυτών των γραφειοκρατικών διαδικασιών γιατί καταργείται η αποστήγη για τα έγγραφα που περιγράφονται, δηλαδή <clears throat> πιστοποιητικά γέννησης, γάμου, πιστοποιητικά εν ζωή, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά κατοικίας, εκλογικά δικαιώματα και απουσία μητρώου. και μπορούν να μεταφραστούν τα έγγραφα αυτά, συνεπώς ε, ε, να εξοικονομήσουν οι ε, πολίτες και τα χρήματα για τους ορκωτούς μεταφραστές. Το σύστημα ανταλλαγής άμεσης πληροφοριών ανάμεσα στις διάφορες δημόσιες αρχές μπορεί να βοηθήσει επίσης. Αν μια υπηρεσία έχει αμφιβολίες για την αυθεντικότητα ενός εγγράφου, μπορεί να έρθει άμεσα σε επαφή με την αρμόδια αρχή σε άλλη χώρα για να επαληθεύσει το αληθές του εγγράφο. Την μέρα που θα δουλέψει πραγματικά η πλατφόρμα αυτή θα βελτιωθεί η ανείχνευση της απάτης πολύ σημαντικά. Η προθεσμία αυτή που προβλέπετε είναι 2,5 χρόνια, είναι μεγάλη, αλλά είναι απαραίτητη έτσι ώστε το σύστημα να τεθεί σε λειτουργία και οι πολίτες να είναι σωστά ενημερωμένοι. Δώσαμε μάχη στο Κοινοβούλιο για να πιέσουμε τις χώρες μέλη και την Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρχει υποχρέωση αποτελεσματικής ενημέρωσης των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να είναι σε γνώση της κατάργησης της αποστήγε όπως επίσης και της ύπαρξης τυποποιημένων πολύγλωσσων εγγράφων το Κοινοβούλιο έδωσε επίσης αγώνα έτσι ώστε το κόστος αυτών των τυποποιημένων εγγράφων των πολύγλωσσων να μην ξεπερνούν το κόστος της απλής μετάφρασης. Τώρα για τη ρήτρα αναθεώρησης, μια έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να αναφερθεί στην περίπτωση αυτή και την πιθανότητα κατάργησης της αποστή για άλλα έγγραφα. Το Κοινοβούλιο ε, είναι ικανοποιημένο εν μέρη μόνο. Θελήσαμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να βάλουμε και άλλα θέματα όπως οι επιχειρήσεις και το νομικό τους καθεστώς. Τα διπλώματα, οι τίτλοι σπουδών, ε, το καθεστώς των αναπήρων. Όλες αυτές οι προτάσεις ε, δυστυχώς δεν έγιναν σε μια πρώτη φάση δεκτές και θα συζητηθούν στα πλαίσια της αναθεώρησης. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα προσέξει να υπάρξει σωστή εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ κυρία Ντελβό. Θα χαιρετήσω τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Τζούροβα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η ελευθερία της ε, κυκλοφορίας δίνει εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρωτοφανείς ευκαιρίες, οι διασυνοριακές προσωπικές και επιχειρησιακές ε, και επιχειρηματικές σχέσεις ανθούν 14 εκατομμύρια πολίτες διαμένουν σε ένα κράτος μέλος, άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής τους. 13% όλων των γάμων στην Ένωση είναι διεθνούς χαρακτήρα και 50% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προβαίνουν σε διασυνοριακές δραστηριότητε, Αναμένω ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Η πρόταση αυτή θα καταστήσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και επιχειρήσεων ευκολότερη, έροντα την γραφειοκρατία. Εδώ είμαστε μετά από τρία χρόνια έντονων διαπραγματεύσεων με τη δική σα αυριανή ψηφοφορία. Η Ένωση θα κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα μπορεί να μην φτάσει στα σέλιδα των εφημερίδων, αλλά πολλοί άνθρωποι θα ανακοφιστούν όταν θα μπει σε λειτουργία, θα τεθεί σε λειτουργία αυτός ο κανονισμός σήμερα. Όταν οι άνθρωποι μετακινούνται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και μετακομίσουν εκεί και θέλουν, χάρη, να αγοράσουν ένα σπίτι, να παντρευτούν ή να κάνουν αίτηση για, για ταυτότητα, εκεί τους ζητούνται, παραδείγματο χάρη, σφραγίδε όπω η σφραγίδα τη Χάγη, επικυρωμένε μεταφράσει. Αυτό είναι εντελώ κάτι που δεν χρειάζεται. Του ζητούνται και ακριβή αντίγραφα βάσει της αρχής της αμοιβέ εμπιστοσύνης ο κανονισμός ε, καταργεί την απέτηση ε, του δημόσια έγγραφα φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης ε, και απλουστεύει τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα επικυρωμένα αντίγραφα και τις μεταφράσεις. Επίσης, εισάγει τα πολύγλωσσα πρότυπα έγγραφα για να αποφευχθούν οι απαιτήσει τη μετάφραση και ενισχύει την καταπολέμηση των ψευδών εγγράφων μέσω τη συνεργασία των κρατών μελών. Το Κοινοβούλιο από την αρχή υποστήριζε αυτόν τον κανονισμό. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμή στον κύριο Ραπκάη, ο οποίο ε, συνέλεξε εύρωστη πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωση στην προηγούμενη θητεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό και του σκιώδει εισηγητέ που διαπραγματεύτηκαν με περισσή ικανότητα ε, τελική το τελικό συμβασμό με το Συμβούλιο. Δεν ήταν εύκολο και έχουμε τώρα ένα ισορροπημένο κείμενο. Καλύπτει ο κανονισμός ε, πολλούς ε, τομείς, πολύ σημαντικούς για τους πολίτες, κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική τους, την εξαρχική τους κατάσταση. Θα είχαμε προτιμήσει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής καθώς και έγγραφα που να είναι χρήσιμα στις επιχειρήσεις να καλύπτονται. Χάρη στην αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου, ο κανονισμός προβλέπει έγκαιρη αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογή. Αυτή η έγκαιρη αναθεώρηση θα επιτρέψει στην Κομισιόν να εξετάσει τη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογή και άλλων τομέων ε, όπως είναι τα θέματα αναπηρίας, ε, τα, τα πτυχία και ε, το καθεστώς εκπροσώπησης των εταιριών. Το Κοινοβούλιο έχει διασφαλίσει επίσης ότι το τέλος που θα χρεώνεται ίσως τους πολίτες για την απόκτηση του πολύγλωσσου εντύπου θα είναι λογικό και τα κράτη-μέλη θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους μέσω των ιστοσελίδων τους και σε επαφές με τους ίδιους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο και τώρα να ακούσουμε τη γνωμοδότηση των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ, ο κύριος Ράντεφ, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Ντελβό, για την έκθεση αυτή. Χάρη στις ε, προσπάθειές της, κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων και σκληρών διαπραγματεύσεων, έχουμε τώρα αυτό το συμβιβαστικό κείμενο σας. Διαβεβαιώ ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, υποχώρησαν, δεν έκαναν εύκολη τη ζωή μας. Γι' αυτό είναι τεράστια η επιτυχία σήμερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι θα καταστήσουμε ακόμη πιο εύκολη την κυκλοφορία των πολιτών και θα πλουστεύσουμε τα δημόσια έγγραφα. Αυτός ο κανονισμός αφορά την άρση των ε, διοικητικών διατυπώσεων όπως είναι παραδείγματο χάρη σφραγίδα της ε, Χάγης και η επικύρωση των εγγράφων εδώ. Αναφερόμαστε παραδείγματο χάρη σε διάφορα έγγραφα, ε, ληξιαρχικά έγγραφα, το ποινικό μητρό κτλ. Επίσης, η διοίκηση στα διάφορα κράτη-μέλη ε, θα μπορεί να επαληθεύει τη γνησιότητα των εγγράφων. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο των πλαστών εγγράφων. Τα πολύγλωσσα πρότυπα έντυπα, τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα θα κάνουν τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη. Θα γλιτώσουν χρόνο στους πολίτες και νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή και να περιλάβουμε και άλλα έγγραφα, παραδείγματο χάρη, που σχετίζονται με τι επιχειρήσει, διάφορα πτυχία, παραδείγματο χάρη πτυχία πανεπιστημίου κτλ. Λυπάμαι που τα κρατημέλη δεν ήταν έτοιμα να δεκτούν τη θέση μα και τώρα όλα αυτά τα έγγραφα δεν ανήκουν στο πεδίο εφαρμογή. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μα εμπιστευτούν περισσότερο την επόμενη φορά που θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε περισσότερα έγγραφα στο πεδίο εφαρμογή και έτσι θα διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο του πολίτε μα. Για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε, 1,5 λεπτό. Κυρία ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πάνω από 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εργάζονται ή σπουδάζουν εκτός ε, ε, των χωρών τους και προσπαθούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Κάθε χρόνο χιλιάδες επίσημα ε, ε, έγγραφα θα πρέπει να σφραγίζονται, να παίρνουν από μια διαδικασία για να αναγνωριστούν στις άλλες χώρες. Θα πρέπει να πλουστευτούν όλες αυτές οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Πρέπει να έχουμε έντυπα σε πολλές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων και εγγράφων που έχουν να κάνουν ε, με την κατοικία τους, με τη διαμονή τους, ε, με την, ε, το λευκό ποινικό μητρό και διάφορες λεξιαρχικές πράξεις και πιστοποιητικά. Αυτό είναι πιο εύκολο λοιπόν για πολίτες που κυκλοφορούν και μετά κομίζουν σε άλλη χώρα. Χαιρόμαστε για τη ρήτρα αναθεώρησης που περιλαμβάνεται στον κανονισμό, η οποία στο μέλλον μπορεί να διευρύνει τον κατάλογο των εγγράφων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ε, ε, άλλα ε, χαρτιά και πιστοποιητικά που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι νέοι κανόνες λοιπόν θα απλουστεύσουν και θα κάνουν πιο εύκολη τη μετακίνηση των πολιτών μας και πολύ σύντομα θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, σαν και 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Ντελβό για τις πολύ δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις και για το ικανοποιητικό αποτέλεσμα που πέτυχε για αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι μόνο ε, έρονται κάποιες διατυπώσεις σχετικά με τα δημόσια εγγραφά που σχετίζονται με το ποινικό μετρό, την κατοικία, την εθνικότητα, αλλά επίσης ε, μειώνεται και το γραφειοκρατικό άχθος που υπάρχει σε πολλές χώρες. Επίσης, είναι καλό νέο ότι δεν χρειάζεται πλέον η σφραγίδα της ε, Χάγης. Εγώ υποστηρίζω και την εισαγωγή αυτών των πολύγνωσων τυποποιημένων εντύπων. Δεν ε, θα χρειάζεται πλέον ε, η σφραγίδα της Χάγης θα μειωθεί και το γραφειοκρατικό κόστος ε, και για τα κράτη-μέλη και θα διευκολυνθούν οι πολίτες στην καθημερινή τους δραστηριότητα και στην κυκλοφορία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό θα διευκολύνει την ε, έκδοση των εγγράφων θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι την εισηγήτρια για την αποτελεσματικότητα με την οποία διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις για τους ε, πρασίνους για 1,5 λεπτό. Κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Δελβό για τη σημαντική της εργασία για την έκθεση αυτή ε, η οποία ήρθε σε αίσιο πέρας. Η αμοιβαία αναγνώριση των δημοσίων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών είναι κάτι το οποίο πραγματικά ε, προάγει και προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία. Αλλά όπως είπε η συγγήτρια, αυτό δυστυχώς ε, ε, εφαρμόζεται για λίγα επίσημα έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλά θα κάνει να κάνει χρήση της ρήτρας αναθεώρησης. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν και άλλα έγγραφα όπως είναι επιστοποιητικά αναπηρίας στον κανονισμό αυτό, διότι όλοι οι Ευρωπαίοι ε, θα πρέπει να χαίρουν όλων των δικαιωμάτων τους παντού με την ελεύθερη κυκλοφορία και ε, οι άνθρωποι με αναπηρίες είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Υπάρχει και μία σύμβαση που επιτέλους για τα άτομα με αναπηρία αύριο αρχίζει και ισχύει στη Φιλανδία, την πατρίδα. Και πολύ θα ήθελα και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η κατηγορία πιστοποιητικών και πρέπει γρήγορα να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που έχουν να κάνουν με την αναπηρία. Good afternoon, everybody. Well, Νομίζω ότι στόχος της ε, νομοθετικής αυτής είναι να διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της απλούστευσης της αποδοχής δημοσίων εγγράφων. Σήμερα λοιπόν κάνουμε το τελευταίο δώρο σε αυτούς οι οποίοι μας απειλούν και οι οποίοι θα κερδίσουν από την πρόταση αυτή μία πρόταση η οποία θα υπονομεύσει ακόμα περισσότερο την εθνική ασφάλεια και θα δημιουργήσει πίεση στα μέτρα ασφαλείας μας. Αυτή η διαδικασία εναρμόνισης λοιπόν αφορά τα έγγραφα τα οποία επιτρέπουν να διακρίνει κανείς, να ξεχωρίζει και να λειτουργεί σαν εμπόδιο σε απειλές. Είναι θα έλεγα αρμοδιότητα των κυβερνήσεων αυτό γιατί αλλιώς δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν από τη λογική της πλήρους ομοιομορφίας. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο φτηνά και ε, αναλώσιμα είναι τα ευρωπαϊκά διαβατήρια. Γιατί εμείς να ε, επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο αυτούς που θέλουν να μας βοηθήσουν. Απορώ για την πρότασή σας. Μου κάνει τρομερή ε, ε, εντύπωση. Ο χρονισμός είναι κακός, ο στόχος είναι κακός και δεν βοηθάει παρά μόνο τους κακούς. Λοιπόν, να το αποσύρετε. Να το αποσύρετε έστω προσωρινά. Και σταματήστε να κάνετε δώρα στους εχθρούς μας. Είναι η άσχημη στιγμή, είναι ο άσχημος τόπος και χρόνος χοντρικά για το INF e 1,5 λεπτό. Κοιτάξτε οι μπλε κάρτες για τις ε, γνωμοδοτήσεις των πολιτικών ομάδων γιατί αυτή τη στιγμή εκφράζονται οι πολιτικές ε, ομάδες και μετά θα ε, αρχίσει ο καθένας να εκφράζεται προσωπικά και θα δεχόμαστε τις μπλε κάρτες. Η κυρία Μπουτονέ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω την προστιθέμενη αξία του εγγράφου αυτού, λόγω ακριβώς των πολλών συμβάσεων που ισχύουν στον τομέα αυτό. Ε, δεν βλέπω το τι συμφέρον έχουμε για αυτά τα πολύγλωσσα κοινά έγγραφα, τα οποία ε, ευτυχώς δεν έχουν καμία αυτόνομη νομική αξία, κάτι το οποίο λυπείται η εισηγήτρια. Το Συμβούλιο έχει μειώσει τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου το οποίο κρατιέται τώρα από τις ρήτρε αναθεώρησης που θέλουν να διευρυνθούν ακόμα οι διαδικασίες διοικητικής διευκόλυνσης. Εγώ νομίζω ότι στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την απάτη και αυτό το έγγραφο δυστυχώς δημιουργεί προβλήματα στις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνε για τον έλεγχο αυτό. Τη στιγμή που διαπιστώνουμε καθημερινά ότι το Σέγγεν είναι επικίνδυνο και ανεύθυνο Τη στιγμή κατά την οποία τα εθνικά κράτη αντιμετωπίζουν μια μεταναστευτική πρόκληση χωρίς προηγούμενο, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκτός κλίματος, προτείνοντας τα ίδια και τα ίδια. Ευχαριστώ. Εδώ τελειώνουν λοιπόν οι πολιτικές ομάδες. Από εδώ και πέρα θα μπορούμε να αποδεχόμεθα τις μπλε κάρτες. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Ζιεύκα, στον κύριο Ζιεύκα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Ευτυχώς έχουμε ομάδες όπως ε, το EFTD και το ε, Εθνικό Μέτωπο στο Κοινοβούλιο που φροντίζουν ε, για την ασφάλειά μας της πατρίδες μας. Ε, ε, έτσι λοιπόν παραμείνετε περίκλειστοι και σας ευχαριστώ που το φροντίζετε αυτό γιατί οι πολίτες της Ευρώπης ξέρουμε ότι περιμένουν κάτι εντελώς διαφορετικό να σας πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το γνωστό επιτέλους το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθετούν νομοθεσία που διευκολύνει την καθημερινή του ζωή. Γιατί αυτός ο κανονισμός διευκολύνει την καθημερινή ζωή εκατομμύριων πολιτών που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μιλάμε για μετανάστες, μιλάμε για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να το αναγνωρίσετε επιτέλους. Αυτός ο κανονισμός έχει ένα πεδίο εφαρμογή που δεν είναι ικανοποιητικό για να είμαι θα πρέπει να είναι ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή, αλλά με κάτι πρέπει να ξεκινήσουμε και οι πολίτες ε, θα μας ευγνωμονούν για, για οποιαδήποτε πράξη διευκολύνει τη ζωή του να μην χρειάζεται να πάνε σε μεταφραστή και να μην χρειάζεται να επικυρώνουν πολλές φορές ε, τα έγγραφα. Ούτε να χρειάζεται να παίρνουν σφραγίδες και υπογραφές ε, στις χώρες ε, όπου μεταβαίνουν. Έτσι λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα θα μας διευκολύνει για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτό το χρόνο. Δεν θα πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή την προσπαθία και θα πρέπει να δούμε πώς θα διευκολύνουμε περαιτέρω τη ζωή, των πολιτών. Παρακαλώ από τον για ένα μισή λεπτό. Ο κ. Σκοφεράτη, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το έργο της κυρίας Δελβό και των σκιωδών εισηγητών είναι εξαιρετικό ο κανονισμός, είναι ένα βήμα προς τα βρός, αν ε, και είναι μετριοπαθής, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Χωρίς αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε τις δυνατότητες που ανοίγονται ενωπιών της. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να πλουστεύουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να μετακινούνται χωρίς τα εμπόδια που συναντούν σήμερα. Όμως δύο πράγματα θα πρέπει να γίνουν επίσης ταχύτατα. Κάτι που, που αναφέρατε εσείς είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να ε, αναγνωρίσουν ε, και να γνωστοποιήσουν αυτή την ομοθεσία γιατί διαφορετικά θα χάσει την αξία της. Εμείς ε, θέλουμε να εφαρμοστεί γρήγορα αυτός ο κανονισμός. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που υπενθυμίστηκε από κάποιον συνάδελφο ο κύριος Βιέφκα, έχουμε περαιτέρω στοιχεία που θα πρέπει να προσθεθούν στον κανονισμό. Σήμερα έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται. Παραδείγματο χάρη έγγραφα που αφορούν τις επιχειρήσεις ε, και έγγραφα που αφορούν και τα άτομα, όπως παραδείγματο χάρη τα πτυχία, ε, τα πιστοποιητικά αναπηρίας, όλα αυτά τα έγγραφα που ουσιαστικά βελτιώνουν την καθημερινή ζωή και σε αυτό χρησιμεύουν και οι νόμοι. Παρακαλώ, κύριε Σκρίπεκ, για ένα λεπτό. Χαίρομαι που κάθε διοικητικό άχθος ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες μειώνεται. Παρ' όλα αυτά ανησυχώ που νέοι ορισμοί και ιδεολογικές αλλαγές μπαίνουν σε, από ό,τι φαίνεται, πρακτικές προτάσεις ε, κυρίως. Ε, εδώ φύγουμε θέματα της οικογένειας και του γάμα. Όμως ε, οι πολίτες ανησυχούν μήπως ε, επιβληθούν πράγματα σε άλλα ε, κράτη, μέλη, παραδείγματος χάρη. Ένα πιστοποιητικό γέννησης παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ταυτότητά τους και τα ονόματα της μητέρας και του πατέρα είναι ιερά θα πρέπει να τα σεβαστούμε όλα αυτά γιατί όλοι μας έχουμε γεννηθεί από ένα πατέρα και μητέρα και έχει δημιουργηθεί μια οικογένεια που είναι πάρα πολύ σημαντική για την δημιουργία των κοινωνιών μας. Σε κάθε κοινωνία χρειάζεσαι πατέρα και μητέρα και αυτό είναι κάτι το πολύ φυσικό. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μακ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Κυρία Γιούροβα, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση στα πλαίσια της δεύτερης ανάγνωσης δεν ψηφίζουμε συνήθως. και ψηφίζεται μια πρόταση παρά μόνο αν κάποιος καταθέσει μια πρόταση άρνησης. Εγώ δεν θα το κάνω και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ υποσχέθηκα στους εκλογείς μου ότι θα καταψήφιζα όλες αυτές τις προτάσεις οι οποίες θα μειώνουν την ελευθερία των πολιτών και πράγματι υπάρχουν μέτρα μείωση της ελευθερίας των πολιτών και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Προβλέπεται ένας ενιαίος τρόπος διατύπωσης επισήμων εγγράφων όπως πιστοποιητικά γέννησης γάμου κτλ. Και αν οι πολίτες μας θέλουν να μεταφερθούν σε μία άλλη χώρα δεν θα χρειάζεται να δίδουν εγκεκριμένες μεταφράσεις κάτι το οποίο καθιστά την έκδοση των εγγράφων αυτών ευκολότερη. Αλλά βέβαια δεν υποχρεώνονται τα κράτη-μέλη να, αποδέχονται τα έγγραφα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να σκεφτώ λίγο περισσότερο και ποιος είναι ο στόχος μας και ο στόχος της Ένωσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ καλό παράδειγμα διακυβερνητικής συνεργασίας. Δεν χρειάζεται να μπλέκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ιστάρα Σφεραγκούτ. Δεν τη βλέπω. Περνάμε τώρα στον επόμενο ομιλητή. Κάουφμαν, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αύριο θα αποφασίσουμε για ένα νόμο που αφορά πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών, άνδρες και γυναίκες, που δεν ζουν στην πατρίδα τους αλλά σε άλλο κρατό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται ή σπουδάζουν. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάνουν χρήση του δικαιώματο στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα χρειαστούν μια ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου, ε, ένα πιστοποιητικό από την αστυνομία, το δίπλωμα οδήγησης ε, γιατί μπορεί να θέλει να γραφτεί στο Δήμο ή ακόμα και να παντρευτεί ή να προχωρήσει σε κάποια άλλη ενέργεια. Μέχρι τώρα δυστυχώς αυτό κοστίζει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα. Ε, έχει φτάσει επιτέλους ο, κόσμο, ο κόμπος το χτένι συγγνώμη, και ε, είναι καλό να καταργηθεί η αποστήλη της Χάγης και ε, να μπορεί ε, ο κόσμος να αποφεύγει την ταλαιπωρία και τις ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες για μια επίσημη μετάφραση. Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω λοιπόν ε, όλους εκείνους τους αδέλφους που είπαν ότι θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Και ε, αυτό να μην αφορά μόνο ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα δηλαδή, αλλά και νομικά πρόσωπα, εταιρείε, όπως αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης και ο κατάλογος των εγγράφων προς αναγνώριση χωράει και άλλα και ποντάρω στη ρήτρα αναθεώρησης γιατί τότε θα έχουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τα πράγματα. Είναι καλό ο νόμος αυτό, αλλά αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα προς τη σωστή επαναλαμβάνω κατεύθυνση δηλαδή προς μια ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την Ευρώπη των δημοσίων εγγράφων. Θα παραμείνω, ε, θα παρακολουθώ το θέμα αυτό όπω και άλλοι συνάδελφοι. Για ένα λεπτό, κύριο Στόμασιτς, παρακαλώ. κυρία Ευχαριστώ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών ε, είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αρθούν όσο δυνατόν περισσότερα διοικητικά εμπόδια που εμποδίζουν τους πολίτες να ζουν και να μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη η Κομισιόν προσπαθεί να προωθήσει την κινητικότητα για να λύσει και το πρόβλημα της ε, ανεργίας. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε όποιον αποφασίσει να μετακινηθεί αλλού. Ούτε η πολιτική ούτε η διοίκηση μπορούν να εμποδίζουν ε, τους πολίτες να λάβουν τέτοιες σημαντικές προσωπικές αποφάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε την ε, χρήση της διοίκησης ε, και τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν αυτές τις διαδικασίες και να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για την κυρία Τόμασιτς. Παρακαλώ. Είπατε ναι, μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι η πρόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης κάποιων επίσημων εγγράφων είναι ένας τρόπος για να διευκολύνουμε, το χάρη, ε, τη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών ή τα ταξίδια. Αλλά, ξέρετε, έχουμε πέντε κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Και αυτοί οι πολίτες έχουν πρόβλημα με την ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν πιστεύετε, παρακαλώ κυρία Τόμας, έτσι να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι τα διοικητικά προβλήματα θα πρέπει να εξαλειφθούν. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στα προβλήματα όσων επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα τους, αλλά και όσοι θέλουν να μείνουν στο κράτος μέλος τους θα πρέπει να τους δώσουμε λόγους για να μπορούν να παραμείνουν. Παρακαλώ η κυρία Κομοντίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η σύγχρονη δημόσια διοίκηση θα διευκολύνει τους πολίτες και θα μειώσει τα γραφειοκρατικά βάρη που είναι ξεπερασμένα. Μιλάμε και για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Το Συμβούλιο όμως από ό,τι φαίνεται δεν συνειδητοποιεί ότι η ψηφιοποίηση θα διευκολύνει τους πολίτες και τις μετακινήσεις τους. Διαρωτώ λοιπόν γιατί ο κανονισμός αυτός αφορά προσωπικά έγγραφα και όχι τους τίτλους σπουδών, τους εκπαιδευτικούς τίτλους. Ε, πολλοί πολίτες είναι αυτοί που χρειάζονται τους τίτλους τους για να μπορέσουν να εγκατασταθούν σε μια άλλη χώρα και υπάρχουν κανονισμοί που καθορίζουν τον τρόπο αναγνώρισης των, των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών τίτλων. Συνεπώς λοιπόν εγώ θα ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν διευκολύνουμε τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται εύκολα τα έγγραφα αυτά. Οι θέσεις του Συμβουλίου δεν μειώνουν τις επιβαρύνσεις της γραφειοκρατικές για τις επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και δεν απλοποιούμε δυστυχώς τη δουλειά των επιχειρήσεων που λειτουργούν διαμεθοριακά. Έπρεπε ο κανονισμός αυτός να μας βοηθήσει να απομακρύνουμε την αχρίαστη γραφειοκρατία. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας, ίσα ίσα τα ψηφιακά μέσα μας επιτρέπουν να είμαστε και αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Ευχαριστώ κύριε Ρέγνερ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Ξέρετε πόσο περίπλοκο είναι ένας Αυστριακός πολίτης, βέβαια θα μπορούσα να φέρω οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ε, να θέλει να περάσει τη σύνταξή του στην ε, Ισπανία και να του πληρώνουν και τη σύνταξη. Θα πρέπει να φέρει ένα πιστοποιητικό ε, ότι ζει ληξιαρχική πράξη η οποία θα πρέπει να ε, μεταφραστεί με ακριβές αντίγραφο και ε, με αποστήλη. Αυτό κοστίζει και ε, χρόνο και χρήμα και θέλουμε να το αλλάξουμε. Η καθημερινή φυσιολογική ζωή στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι απλή. Οπότε μέσω και μακροπρόχρονα χρειάζεται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό επίσημο έγγραφο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα πιο μετριοπαθές αποτέλεσμα από εκείνο που θα ήθελε η κυρία Ντελβό αλλά και σκιώδης ηγητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχικά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι έχει γίνει αυτό το βήμα. Τώρα ε, θα επωφεληθούν οι πολίτες, καταργείται η αποστήλη για ε, ορισμένα δημόσια έγγραφα, όπως είναι η πράξη γέννησης και θανάτου. Και επιπλέον πολλοί νέοι ε, ενήλικοι ε, πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Παραμένει λοιπόν προτεραιότητα για μας να τους διευκολύνουμε τη ζωή και να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση ε, απολυτηρίων λυκείου και διπλωμάτων της δευτεροφάθμιας εκπαίδευσης. Ας είναι λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα. Το θέμα αυτό θα το παρακολουθούμε γιατί θα συμβάλλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Εύελιν. Svoboda για 1,5 λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό, την εισηγήτριά μας και όλους όσους πήραν μέρος στην κοινή αυτή προσπάθεια. Τους ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειες που έκαναν. Η συμβιβαστική πρόταση αποδεικνύει τις πραγματικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Συνειδητοποιώ ότι ο, εμπιστο, ο εμπιστευτικός χαρακτήρας ορισμένων εγγράφων και η εμπιστοσύνη καλύτερα στα έγγραφα αυτά βοηθούν την κοινωνία να λειτουργήσει και γι' αυτό ό,τι αλλάζει τους κανόνες πρέπει να είναι πάρα πολύ σταθμισμένο. Όμως νομίζω ότι οι πολίτες ε, περιμένουν περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι απλά μια αργή και σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα. Ε, λυπάμαι που τα κράτη-μέλη δεν θέλησαν να προχωρήσουν περαιτέρω. Τουλάχιστον όπως είχε προτείνει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, Περιορίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά κάποιες περιπλοκές, αλλά ας ξεκινήσουμε τη δημιουργία ενός πραγματικού κοινού χώρου. Μόνο ένα τέτοιο μέτρο θα επηρεάσει και τους πολίτες, τους απλούς και τους επιχειρηματίες. Παρακαλώ για μισή λεπτό, κύριο Τσάκη. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια πολίτες ε, που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν διαμένουν σε ένα ολοκληρωτός μέλος ε, πρέπει οι πολίτες να αντιμετωπίσουν άγνωστα εκπαιδευτικά, φορολογικά και άλλα συστήματα. Έτσι λοιπόν τίθεται διοικητικά προβλήματα. Απλουστεύοντας τις διαδικασίες, αυτός ο κανονισμός επικεντρώνεται στην διασυνοριακή αποδοχή των δημοσίων ε, εγγράφων, των λεξιορχικών εγγράφων. Έτσι λοιπόν χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία καθώς έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που επικυρώνονται κάθε χρόνο παγίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών θα επιτρέψει στους πολίτες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Ε, πραγματικό πλεονέκτημα του κανονισμού είναι ότι εισάγονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ε, ουσιαστικά παραδείγματος χάρη ε, ευνοεί ε, τις κοινότητες που είναι εγκατεστημένες σε κάποιες χώρες και μιλούν μια άλλη γλώσσα. Αυτός ο κανονισμός είναι λοιπόν καλό σημείο φετηρίας και θα ήθελα να τον υποστηρίξω. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς επιτρέψτε μου και μένα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους και ηγητές για την έκθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζεται βασικά από τις ελευθερίες, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, ε, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ε, ε, ισχύει η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων παρά το γεγονό ότι δίνουν όλα τα κράτη-μέλη και μέλη του Σέγγεν. Δυστυχώ όμω υπάρχει αυτό το γραφειοκρατικό άχθο στη διασυνοριακή αποδοχή ε, επισήμων εγγράφων και αυτό επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε και άλλα πρακτικά εργαλεία έτσι ώστε να απλουστεύεται η ζωή των πολιτών μας όταν ταξιδεύουν εκτός των συνόρων τους. Η ε, ενότητα ε, και η διαφορετικότητα θα πρέπει να βρίσκουν έκφραση και στη γραφειοκρατία και στο δημόσιο οι πολίτες έχουν ε, καινούργιες ανάγκες και νέες επιθυμίες ε, και ε, αγωνιούν για μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα την κατάσταση. Ας είναι αυτό ένα πρώτο βήμα σε ένα πιο στενό επίπεδο. Τα πιστοποιητικά για την οικογενειακή κατάσταση ελπίζω στο μέλλον να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η αρχή της ε, ε, ε, ασφάλειας δικαίου, της γνησιότητας των εγγράφων και δεν θα πρέπει να μας παρασύρει αυτή η οπτασία της ελεύθερης κυκλοφορίας και της απλούστευσης. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ταμπαρντέλ, έχεις το λόγο ένα λεπτό. Αγαπητέ Επίτροπε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων που ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα από τη χώρα προέλευσης. Η πρόταση απλούστευσης της διαδικασίας αποδοχής δημοσίων εγγράφων είναι πολύ σημαντικό και για τους πολίτες και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οι τουρίστες και οι εργοδότες που πρέπει να αποδείξουν ότι πληρώνουν στους φόρους τους, οι φοιτητέ που έχουν σχέσεις με τα πανεπιστήμια τους, η γραφειοκρατία είναι εμπόδιο στην ελευθερία και γι' αυτό η πρόταση της Επιτροπής είναι απαραίτητο βήμα αλλά όχι επαρκές. Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου έχουν αυξήσει τον αριθμό των εγγράφων που γίνονται αποδεκτά από τις εθνικές αρχές και μεταφέρουν κάποιες από τις ευθύνες από τους πολίτες στις αρχές. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και λιγότερο χρόνο να ξοδεύουν όπως και λιγότερα χρήματα. Είναι μια καλή πρωτοβουλία, είναι μια πρωτοβουλία που θα βελτιώσει το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη και τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς, ένα λεπτό είναι ιδιαίτερα οξύμορο τη στιγμή που πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν αναστείλει τη Σέγγεν να συζητούμε την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της άπης ορισμένων εγγράφων. Φυσικά η διευκόλυνση των πολιτών είναι κάτι σημαντικό και αυτό θα γίνει με την κατάργηση της σφραγίδας αποστήλ. Πρόκειται για θετικό γεγονός που θα ενισχύσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, την εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες και την ανέβρεση εργασία όμω θα πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των δημοσίων εγγράφων και ιδίως αυτά που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε τα θέματα ασφάλειας τα οποία τέθηκαν. η ανάγκη της αναγνώρισης των εγγράφων και της κατάργησης της αποστήλη είναι επίκαιρη ιδίως τώρα που έχουμε μεγάλη μετανάστευση των νέων από τις χώρες του νότου και ιδίως από την ελλάδα καθώς χιλιάδες επιστήμονες έχουν πάει πλέον στις χώρες του βορρά. πρόκειται για ένα brain drain για μια αφέμαξη εγκεφάλων που πρέπει να σταματήσει και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πέραν από την διευκόλυνση θα πρέπει να δούμε και με μέτρα για τη στήριξη της ευρωπαϊκής περιφέρειας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αυτή η πρόταση είναι υπέρ των πολιτών και υπέρ της εσωτερικής αγοράς. Έχει απόλυτο νόημα να έχουμε ενιαία έγγραφα σε πολλές γλώσσες. Ε, καλωσορίζω αυτό το κανονισμό ως πρακτικό παράδειγμα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται προς όφελος των ε, κανονικών πολιτών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έχει να κάνει με τα πιστοποιητικά και τις λεξιαρχικές πράξεις ε, γέννησης, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα για τις επίσημες μεταφράσεις διπλωμάτων και τίτλων σπουδών. 6 με 8% γνωρίζουμε των πολιτών τη ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν σε άλλα κράτη-μέλη. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ε, ότι η ε, κυκλοφορία αυτή θα πρέπει να γίνεται όσο ε, γίνεται πιο απρόσκοπτα. Ιδιαίτερα για τους Ιρλανδούς αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί τους ζητούν πάρα πολλά έγγραφα. Ε, το γεγονό λοιπόν ότι θα έχουμε στάνταρ τυποποιημένα έγγραφα σε πολλέ γλώσσε είναι πάρα πολύ εύστοχο. Θα πρέπει να είμαστε όμω και τολμηροί αλλά και φιλόδοξοι για το μέλλον. Γι' αυτό το βλέπω ω ένα μόνο βήμα και το πρώτο και όχι το τελευταίο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που προφέρετε σωστά το όνομά μου. Γιατί συνήθω είναι πολύπλοκο να το προφέρει κανεί. <laughs> ακόμη και για τους Ιταλούς. Έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα που έχει αρχίσει να λειτουργεί στην Κροατία και λειτουργεί πάρα πολύ καλά και θα πρέπει να μας καθοδηγήσει μέσω του συστήματος e-Citizen, ηλεκτρονικός πολίτης, ε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχουν οι πολίτες. Ας ξεκινήσουμε από αυτά τα κυρία έγγραφα, αλλά μην σταματήσουμε εκεί. Ας πάμε παραπέρα. Ας συμπεριλάβουμε τους τίτλους, τα πτυχία, όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για την απασχόληση, όλα όσα χρειάζονται οι πολίτες. Ας μην σταματήσουμε εδώ, ας προχωρήσουμε. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητή για ένα λεπτό. Η απαλλαγή από την υποχρέωση επικύρωση και επισημείωση συγκεκριμένων δημοσίων εγγράφων αποτελεί σημαντικό βήμα προ τον περιορισμό τη γραφειοκρατία και τη μείωση τη ταλαιπωρία των πολιτών τη Ένωση. Δημόσια έγγραφα τα οποία δύναται να αναζητηθούν γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών και να πιστοποιηθεί η γνησιότητά του σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδι στι επαγγελματικέ ακαδημαϊκέ και προσωπική φύσεω δραστηριότητε των ευρωπαίων πολιτών. τρόποι μέθοδοι και τεχνικέ υπάρχουν και συνεχώ βελτιώνονται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. τα κράτη μέλη οφείλουν να ξεφύγουν από τι όποιε τυχόν αγκυλώσει τα συγκρατούν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωή των πολιτών του περιορίζοντα την άσκοπη και οικονομικά ζημιογόνα ταλαιπωρία σε τέτοιου είδου διαδικαστικά θέματα το πεδίο εφαρμογή των συγκεκριμένων διοικητικών διευκολύνσεων είναι ακόμη περιορισμένο αλλά δύναται και οφείλει να επεκταθεί και σε άλλα έγγραφα όχι όμω ει βάρο τη αξιοπιστία και τη ασφάλεια των εγγράφων. ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση του κυρίου Ναγκρέσκου. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα που έγινε με το νέο κανονισμό που καταργεί την υποχρεωτική ε, σφραγίδα αποστηλή για ε, τέτοια έγγραφα όπως είναι η εθνικότητα, η διαμονή, το ποινικό μητρό. Ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε ενιαία έντυπα σε πολλές γλώσσες. Έχω όμως και επικρίσεις. Πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω γιατί ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει ε, τίτλους σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης, πτυχία, ε, πιστοποιητικά αναπηρίας και δεν συμμαζεύεται. Ε, δεν κατάλαβα, οι φοιτητέ, οι επιχειρηματίε, τα άτομα με αναπηρία δεν δικαιούνται να ταξιδεύουν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται και τόσο χρόνο για να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Για ποιο λόγο, μία τριετία για να ε, εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ε, ηλεκτρονικό για να τσεκάρουμε τα έγγραφα και γιατί να κοστίζει περισσότερο η επιστοποίηση τη γνησιότητα. Εγώ ζω στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και τα αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα και είναι εκατομμύρια οι Ρουμάνοι που ζουν εκτό των συνόρων. Ε, και ευχαριστώ και παρακαλώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν κι άλλο. Μάλιστα, για τις απαντήσεις τώρα η κυρία Γιούροβα, καταρχήν και κατόπιν η Παρακαλώ, η Επίτροπος. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ο συμβιβασμός ε, στον οποίο φτάσατε με το Συμβούλιο θα φέρει από τα ωφέλη στους πολίτες μας και δεν θα χρειάζεται πλέον να ξοδεύουν χρόνο και χρήμα προκειμένου να σφραγιστούν τα εγγραφά τους από μια δεύτερη αρχή στο κράτος μέλος τους πριν να μπορέσουν να τα παρουσιάσουν στην αρχή ενός άλλου κράτους μέλους. Και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι και εγώ το κατανοώ αυτό σε ένα πρωτοβήμα σε μια μακροπρόθεσμη διαδρομή και ορθώς είπατε ότι πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω και μπορώ να σας πω ότι έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδρομή πριν 7 χρόνια όταν είχαμε σχεδιάσει ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τους πολίτες μας που ταξιδεύουν και θέλουν να μετικήσουν σε άλλο κρατός μέλος. εφαρμόζοντα ε, το δικαίωμα, απολαμβάνοντα το δικαίωμα τη ελεύθερη μετακίνηση, τη ελεύθερη κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού για να εργαστούμε περαιτέρω επί του ζητήματος και άκουσα αναφερθήκατε στα ε, πτυχία, στα έγγραφα που σχετίζονται με τα πιστοποιητικά αναπηρία, στα έγγραφα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Θέλουμε φυσικά και οι επιχειρήσεις να υποφεληθούν αυτού του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα φυσικά και ανυπομονώ να συνεργαστώ περαιτέρω μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ντελβό, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την υποστήριξή τους, την σύνδρομή τους. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε ίσως ε, ε, να διασώσουμε ε, κάποιες προτάσεις στις οποίες στην πρώτη ανάγνωση είχαν τύχει πλειοψηφίας. Καταρχάς θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ένα συγκεκριμένο βήμα αν και ε, θα έλεγα σχετικά περιορισμένο. Δεύτερον, η πλατφόρμα αυτή η οποία δημιουργεί το δίκτυο ανάμεσα στις δημόσιες διοικήσεις και επιτρέπει την άμεση ανταλλαγή στοιχείων αντίθετα με αυτά τα οποία υπόθηκαν από ορισμένου, είναι εξαιρετικό μέσο καταπολέμησης της απάτης και θα επιτρέψει την κατάργηση ε, της χρήσης μιας φραγίδας της οποίας πολλές φορές αμφισβητείται η αυθεντικότητα, η γνησιότητα. Η πρόταση αυτή, ο κανονισμός αυτός θα είναι ένα σημαντικό βήμα εφόσον ενισχύσει την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχουμε ανάγκη από την εμπιστοσύνη αυτή αν πράγματι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο και να κινητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Και τέλος, σας μου επιτρέψετε, Επίτροπε, να πω ότι δεν εγκαταλείπω την ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μπροστά μας μία πρόταση η οποία θα επιτρέψει όχι μόνο την αποδοχή των δημοσίων εγγράφων, αλλά και την αυτόματη αναγνώρισή τους και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Μάντι, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Πάλι η έκθεση της κυρίας Ντελβό για τη μεταβίβαση